Sí. Buenas tardes. Καλό σας απόγευμα. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας με το σημείο 12. Προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας σε σχέση με τον κανονισμό για το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ιώσιπ Βιλαβέρ, τον Υπουργό Θαλάσσης ε, Μεταφορών και Υποδομών, που είναι και το υπεύθυνο Υπουργείο στην Κροατία για το συγκεκριμένο κανονισμό. Μιλάμε λοιπόν για τον κανονισμό ε, που έχει να κάνει με την ιδιωτική ζωή σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Το Υπουργείο λοιπόν Θαλάσσιων Μεταφορών και Υποδομών είναι η αρμόδια αρχή για το θέμα αυτό, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικών ασχολούνται με τους άλλους φακέλους που έχουν να κάνουν με την προστασία δεδομένων και θα έρθουν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την ερχόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε του λοιπούς φακέλου που έχουν να κάνουν με την προστασία δεδομένων. Η πρόταση κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ε, ηλεκτρονικά ε, είχε υποβληθεί το 2017. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πήρε θέση τον Οκτώβριο του 2017 επί του κειμένου που εγκρίθηκε στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Στο Συμβούλιο, συγκεκριμένο φάκελο, για να περιπλέξουμε ακόμα λίγο τα πράγματα, εξετάζεται στην ομάδα εργασία τηλεπικοινωνιών. Που δεν αποτελείται από του ίδιου εκπροσώπου των κρατών μελών που ασχολούνται με το GDPR. Έτσι λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Διάφορες προεδρίες ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία για αυτή την πρόταση επιφυλακτικής Προεδρίας το προηγούμενο εξάμεινο. Η νέα Προεδρία, η Κροατική Προεδρία λοιπόν, ήρθε να μας παρουσιάσει τις δικές προτεραιότητες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας σε Κάμπος Μπορδόν ε, εξέδωσε μία απόφαση πρόσφατα ε, σημαντική ε, για το ζήτημα αυτό, την παρακράτηση δεδομένων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπιλαβέρ που είστε εδώ μαζί μας. Έχετε τον λόγο, είναι τιμή μας που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Στη συνέχεια θα δούμε ποιες πληροφορίες θα προκύψουν ε, ποιε ερωτήσει μόνο θα προκύψουν από τα μέλη. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή. Καλό απόγευμα σε όλου. Σα ευχαριστώ όλου που ήρθατε και που επιδείξατε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Είναι τιμή μου που μιλώ εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο όνομα του Κροατικού Υπουργείου Θαλάσσιων Μεταφορών και ε, υποδομών και εκ μέρου του Συμβουλίου βεβαίω. Θα αναφερθώ στο σκέλος του προγράμματος της Κροατικής Προεδρίας που έχει να κάνει με την τηλεπικοινωνία και την κοινωνία της πληροφορίας και που σχετίζεται με αυτή την επιτροπή. Το όνομά μου είναι Γιώση Μπιλάβερ, είμαι υφυπουργό ε, στο Υπουργείο Θαλάσσης Μεταφορών και Υποδομών, υπεύθυνο και για τα ζητήματα τηλεπικοινωνιών. Ε, η παρουσίασή μου και η παρουσίαση των προ, προ, μας ε, ε, την έχω προετοιμάσει στη δική μου γλώσσα, στα κροατικά και θα συνεχίσω στη γλώσσα αυτή την παρουσίαση. Κυρίε και κύριοι, όπως γνωρίζετε, η Κροατική Προεδρία ανέλαβε τα καθήκοντά της ε, σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για την Ένωση καθώς αρχίζει ο νέος θεσμικός κύκλος και νομοθετικός κύκλος. Το πρόγραμμα της Κροατικής Προεδρίας βασίζεται σε τέσσερις προτεραιότητες με βάση τις κατές γραμμές ε, τη νέα στρατηγική ατζέντα του Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2024 και σύμφωνα και με το πρόγραμμα του τρίο των Προεδριών Ρουμανία, Φιλανδία και Κροατία. Το σλόγγαν της Προεδρίας μας είναι μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Τέσσερι είναι βασικέ προτεραιότητες, όπως είπα. Μια Ευρώπη που αναπτύσσεται, μια Ευρώπη που συνδέεται, μια Ευρώπη που προστατεύει, μια Ευρώπη που επηρεάζει. Σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε αυτή τη Επιτροπή, η Ευρώπη που προστατεύει του πολίτε τη είναι μια σημαντική προτεραιότητα, όπω αντιλαμβάνεστε, και ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η σχετική προτεραιότητα είναι η Ευρώπη που συνδέει. Σε ό,τι αφορά τώρα το αντικείμενο της παρουσίασής μου έχει να κάνει με τον κανονισμό σχετικά με την τρονική ιδιωτική ζωή ε, είναι βασικό ε, στοιχείο για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς όπως θα ακούσατε και στην εισαγωγή αρχικά ο κανονισμός αυτός ε, ήταν να τεθεί σε ισχύ από κοινού με το GDPR δυστυχώς όμως αυτό δεν συνέβη τελικά η πρόταση κανονισμού αυτή έχει παραμείνει στην νομοθετική διαδικασία ακόμα εκρεμή ενώ το GDPR εφαρμόζεται ήδη εδώ και κάποιο καιρό. Είναι η έβδομη συνεχόμενη προεδρία η δική μας ε, η οποία προσπαθεί να σημειώσει πρόοδο. Οι προκάτοχοί μας έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε συμβιβασμό έτσι ώστε η νομοθετική διαδικασία να προχωρήσει και οι διαπραγματεύσει, οι διαθεσμικές ε, να μπορέσουν να τελεσφορήσουν. Ε, θέλω να υπογραμμίσω τις προσπάθειες που έχει κάνει η Φιλανδική Προεδρία ε, που προσπάθησε να φτάσει σε γενική προσέγγιση γύρω από ένα συμβαστικό κείμενο. Τελικά όμως η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή σε επίπεδο κορεπέρ. Και αυτό μα οδήγησε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να ανοίξουμε ξανά τι συζητήσει για όλα τα εκκρεμή ζητήματα και να φτάσουμε ε, σε συμφωνία. Δεν είναι εύκολα τα θέματα αυτά δυστυχώς. Ε, πρόκειται και κάποια πολύ ουσιαστικά στοιχεία ε, της πρότασης, η σχέση με το GDPR, ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ του πεδίου εφαρμογής του GDPR και του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού. Επιπλέον, και υπάρχουν και άλλα εκρεμή ζητήματα, τα στοιχεία της επεξεργασίας δεδομένων, οι στόχοι μάλλον, οι, οι λόγοι ε, ε, το θέμα των cookies που επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη ε, σε ιστοσελίδες, ε, επίσης θεσμικές διατάξεις ώστε να μπορούν διάφορα εθνικά ε, όργανα να είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του κανονισμού. Υπήρχαν και στοιχεία που δεν, ήταν, δεν αποτελούσαν μέρο τη αρχική πρόταση, αλλά που προέκυψαν στη συζήτηση η καταπολέμηση του περιεχομένου που περιλαμβάνει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ε, επίσης, ε, η κοινοποίηση σχετικά με την παρακράτηση δεδομένων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν είναι λοιπόν εύκολα όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι πολλά τα εμπόδια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια του κανονισμού αυτού για την e-privacy. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Είμαι πεπισμένος ότι ο στόχος είναι κοινό για όλους να έχουμε δηλαδή ένα κανονισμό που θα επιτρέπει να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας ε, των συμπολιτών μας και της ιδιωτικής ζωής τους και βεβαίως πρέπει και ο κλάδος να έχει το απαραίτητο περιθώριο για να εξελιχθεί, για να καινοτομήσει. Ε, εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσουμε τη συνδεσιμότητα και να θεσπίσουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά. Η ανάπτυξη των δικτύων 5G είναι άλλη μία από τι προτεραιότητέ μα. Θεωρούμε ότι τα συμπέρασματα του Συμβουλίου επί Προεδρία ε, είναι κρίσιμα για το ζήτημα αυτό. Θα φροντίσουμε να εφαρμοστούν. Υπάρχουν και άλλε ζητήματα όπω η τεχνητή νοημοσύνη. Αναμένουμε την σχετική πρόσθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πάρει τη μορφή λευκή βίβλου από όσο ξέρουμε. Σκοπεύουμε να συζητήσουμε το κείμενο αυτό έτσι ώστε η μελλοντική νομοθεσία να ακολουθήσει τον τη σωστή οδό. Θα φροντίσουμε όλες οι δραστηριότητες μας προφανώς να συνδέονται, να, να, να ευθυγραμμίζονται μάλλον και με το Green Deal και ε, βεβαίως ε, η οικονομία να είναι ουδέτερη σε ό,τι κλιματική ε, επίπτωση. Ευχαριστώ πολύ, ήσασταν σύντομος και περιεκτικός. Είναι εδώ και η εισηγήτρια αυτού του σημαντικού φακέλου που είναι η κυρία Ζήφελ και θα της δώσουμε το λόγο και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στους ε, υπόλοιπους ε, συναδέλφους που είναι σκιώδεις εισηγητές. Καταρχήν, η κυρία Ζήπελ ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Κρότικη Προεδρία για την παρουσίαση αυτή. Θα πρέπει να αναφερθώ σε κάποιες συζητήσεις που είχαμε σήμερα το πρωί. Οπότε το Κοινοβούλιο κατηγορήθηκε όταν συζητήσαμε το θέμα των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων ε, ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο online ότι μπλοκάρουμε τις εργασίες και καθυστερούμε. Όμως κάνουμε τη δουλειά μας. Ε, από την άλλη, ποτέ δεν άκουσα, ιδίως από την Κομισιόν, ε, κάποια κριτική απέναντι στο Συμβούλιο γιατί αυτή είναι υπερβολικά βραδής Και αυτή δεν αποτελεί κριτική στην Κροατική Προεδρία, αλλά στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο στο σύνολό του. Γιατί, αν σας κατάλαβα καλά, είπατε τώρα ότι πρόκειται τώρα ήδη για την 7η Προεδρία που ασχολείται σε κάποιο βαθμό με το e-privacy και εξακολουθούμε να μην έχουμε λύσεις και απαντήσεις. Επίσης, ορθώς είπατε, ότι όταν ε, λαμβάνουμε αποφάσεις ή παρουσιάστηκε αυτός ο φάκελος, ε, θα θεωρήσει η Κομισιόν ότι είναι μικρή αδελφή του GDPR, του Ελληνικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων. Έτσι λοιπόν πολύ εύκολα θα μπορούσε να προσθεθεί στους κανόνες του GDPR και έχουμε δύο λόγους ε, για τους οποίους έγινε αυτό. Καταρχήν η υφιστάμενη οδηγία για το e-privacy εφαρμόστηκε με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Πολύ συχνά δεν εφαρμόστηκε ορθά. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ζητήσαμε κανονισμό. Ο άλλος λόγος ήταν ότι η οδηγία δεν είναι πλέον επικαιροποιημένη. Παραδείγματο χάρη, υπήρξε ανάγκη να δημιουργηθούν ίσοι κανόνε για όλου ε, του πρωταγωνιστέ ε, και για τι εταιρείε τηλεπικοινωνιών, αλλά και για όλε τι υπηρεσίε ε, over the top. Αυτή ήταν η υποκείμενη ιδέα και η ευρύτερη η ιδέα ήταν ότι πέρα από το GDPR θα πρέπει να προστατεύσουμε και την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών ως θεμελιώδες δικαίωμα. Επομένως, ε, είναι ανησυχητικό ότι τα κράτη-μέλη δεν σημειώνουν πρόοδο σε αυτό το βαθμό και αντί να επικεντρωνόμαστε στα κύρια στοιχεία του e-privacy, το Συμβούλιο εισάγει νέες πτυχές για να δυσκολέψει ακόμη περισσότερα τα πράγματα. Παραδείγματο χάρη στι συζητήσει που αφορούν τη διατήρηση των δεδομένων. Λυπάμαι. Αν θέλετε να έχετε διατήρηση των δεδομένων, το θέλετε κρατημένο, να δημιουργήσετε ένα νέο νόμο. Ζήτηστε την Κομισιόν να δημιουργήσει νέο νόμο, αλλά δεν μπορείτε αυτό να το κάνετε μέσω του φακέλου μιας άλλης νομοθεσίας. Επίσης ακούσαμε ότι κάποια κράτη-μέλη θέλουν εξαιρέσει από το δικαίωμα ε, για να προστατεύσουν την ε, εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και λένε όταν μιλάμε για τη σεξουαλική καταπίεση υποδιών και την παιδική πορτογραφία πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση. Και πάλι, συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό αδίκημα και θα πρέπει να εργαστούμε από αυτού. Δεν μπορείτε όμω ε, να έχετε την εξαίρεση αυτή σε μια νομοθεσία όπου ακριβώ λέτε πρέπει να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών. Αν έχετε ένα συγκεκριμένο φάκελο και έχετε αποδείξει ότι κάποιο συνδέεται με ένα τέτοιο αδίκημα ή με κάποιο άλλο αδίκημα, τότε έχουμε διαδικασίε σε όλα τα κράτη-μέλη και στην Ευρώπη για να ληφθεί απόφαση από τον εισαγγελέα ή τον δικαστή και να αποφασίσεις στη συγκεκριμένη ε, περίπτωση δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το privacy αλλά ε, μπορείς να έχεις ε, μια γενική εξαίρεση σε έναν φάκελο ε, που μιλά για την εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας. Τώρα, βεβαίως ε, θα ήθελα να έχουμε απόφαση από το Συμβούλιο, πέρα από την κριτική που ανέφερα, για να μπορέσουμε επιτέλους να ξεκινήσουμε τους τριμμένους διαλόγους για αυτή τη σημαντική υπόθεση. Αλλά αν η Κομισιόν δεν είναι πρόθυμη να το πράξει αυτό, ίσως μπορεί να το ζητήσει το Συμβούλιο. Γιατί σε κάποιε περιπτώσει ήδη είχαμε αποφάσει όπου οι αρχέ προστασία των δεδομένων και άλλε αρχέ βρήκαν ότι σε συνδυασμό με την οδηγία για την ψηφιακή ιδιωτικότητα και τον Γενικό Κανονισμό Προστασία των Δεδομένων, κάποια πράγματα είναι παράνομα και άρχισαν διαδικασίε επί παραβάση. Και αν η Κομισιόν δεν είναι πρόθυμη να ξεκινήσει τι ανάλογε διαδικασίε, ίσω θα μπορούσε το Συμβούλιο να επιληφθεί και τελικά τα κράτη-μέλη ίσως να είναι πιο έτοιμα να πούν εντάξει τελικά θα παρουσιάσουμε μια απόφαση για το e-privacy για την ψηφιακή ιδιωτικότητα παρά να βλέπουμε περισσότερες διαδικασίες επί παραβάση. Ίσως λοιπόν μπορούμε να σκίσουμε πίεση σε κάποια κράτη-μέλη που δεν θέλουν να πάνε παραπέρα. Ευχαριστώ κύριε Σίπελ. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας ως εισηγήτρια. Κυρία Ιντβελτ, εξ ονόματος του Ρινιού, να θέλει το λόγο σκιώδης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομη. Καταρχήν, συμφωνώ με την εισηγήτρια και όσα είπε. Είναι πολύ ενοχλητικό ότι περιμένουμε για πάνω από δύο χρόνια. Νομίζω ότι το Δεκέμβριο του 2017 Διαθετήσαμε την πράξη αυτή και αν το Συμβούλιο κάνει μια καθολική δουλειά, είμαι ευχαριστημένη. Εδώ ε, αυτό είναι γελίο. Είναι ένα από του τομεί όπου δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του Συμβούλιο ω νομοθέτη. Και η Ευρωπαϊκή, Κομισιό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ελπίζω να μα ακούει, τότε ε, όταν δεν μπορεί να συμφωνήσει το Συμβούλιο, σκέφτεται μήπως να αποσύρει κάποια πρόταση αλλά επειδή το Συμβούλιο δεν κάνει τη δουλειά του, δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να καταχράτει την εξουσία της όταν οι άλλοι έχουν κάνει τη δουλειά τους, οι άλλοι νομοθέτες. Θα ήθελα να μάθω και επί της ουσίας τι θέματα συζητούνται, αλλά και τι πλειοψηφίε θα είχατε στο Συμβούλιο. Γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχει μια τάση στο Συμβούλιο να αρνούνται να εφαρμόσουν τη Σύνδεξη Λισαβόνας και να περιμένουν για πλήρη ομοφωνία. Καθώς το Κοινοβούλιο θέτησε τη θέση του, το 17, πολλά έχουν γίνει στον κόσμο και ξέρουμε πολλά περισσότερα για τους τρόπους που χρησιμοποιούνται και υπάρχει κατάχρηση των δεδομένων για να υποσκάψουν τις δημοκρατικές μας εκλογές. Παραδείγματος χάρη είδαμε τι έγινε με την Cambridge Analytica και κάποιες άλλες εξελίξεις. Ακόμη και αν το Κοινοβούλιο λοιπόν θέτει σε μια θέση που προβλέπει πολύ ισχυρή προστασία Νομίζω ότι ούτε καν εμεί υποψιαζόμασταν αυτέ τι εξελίξει που θα λάμβαναν χώρα ακόμη και μέσα σε δύο χρόνια μετά την οθέτηση από το Κοινοβούλιο, που ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τη θέση μα. Ελπίζω λοιπόν ότι οι υπουργοί στο Συμβούλιο επίσης συνδετοποιούν το τι συμβαίνει παγκοσμίω και το υιοθετήσουν. κάτι η πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία των πολιτών, αλλά και η προστασία των κοινωνιών μας και της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νετφέλτ. Από τους Πρασίνους και την Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία, το λόγο έχει ο κύριος Μπράιερ. Παρακαλώ. Thank you, Chair. As my... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε ένα νομικό εργαλείο για την ε, ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο. Γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών. Αυτό δεν λύνεται με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, αλλιώς δεν θα χρειαζόταν τίποτα άλλο. Οι ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες είναι πάρα πολύ ευάλωτε στις υποκλοπές και χρειάζονται ιδιαίτερη ε, προστασία. Υπάρχουν τα λεγόμενα μεταδεδομένα για τις επαφές που έχουμε, για τη χρήση του ίντερνετ, για τις μετακινήσεις μας. Αυτό συστηματικά συλλέγεται και είναι αντικείμενο εκμετάλλευση σε μεγάλη κλίμακα. Ε, υπάρχει η ε, προστασία των δεδομένων, των πηγών, των δημοσιογράφων. Υπάρχουν θέματα χειραγώγησης της κοινή γνώμη. Και τι θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες από τη συλλογή και εκμετάλλευση τέτοιων μεταδεδομένων. Για να μην ε, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού, ανείχνευσης και, και καλά μιλήσατε και για το κλίμα και για το περιβάλλον, αυτό είναι μια άλλη πτυχή και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά αυτό που συζητάει το Συμβούλιο είναι το αντίθετο. Είναι μαζική αποδυνάμωση αυτού που ισχύει τώρα στην οδηγία για το ηλεκτρονικό απόρριτο. Δηλαδή θέλουν ακόμα μεγαλύτερη μαζική ε, συλλογή χίδιν έτσι στοιχείων και δεδομένων. Ξέρω ότι μαζικά έχετε δεχτεί πιέσεις από την ε, βιομηχανία και τις διαφημιστικές εταιρείες κυρίως και υπάρχουν ε, και κάποιες διατάξεις που σχεδιάζεται ε, για το φιλτράρισμα και ε, τη λογοκρισία. Φανταστείτε να σας ανοίγει το ταχυδρομείο τα γράμματά σας την ιδιωτική αλληλογραφία για να ελέγχει μήπως υπάρχει κανένα αθέμητο μήνυμα. Μα γίνονται τέτοια πράγματα στη δημοκρατία, αν σας ανοίγουν την ιδιωτική αλληλογραφία. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να ζω σε τέτοια κοινωνία. Και αυτό έχει να κάνει και με ένα άλλο που συζητήσαμε, ε, γιατί αυτό ανοίγει την πόρτα για μαζική ε, αποθήκευση και κράτηση δεδομένων. Για κάθε τηλεφώνημα, για κάθε ε, σύνδεση με το διαδίκτυο, κάθε πολίτη, συλλογικά για τον πληθυσμό. Είναι τεράστια συλλογή δεδομένων μαζικής κλίμακας που παραβιάζει με τρόπο κατάφορο και δυσανάλογο ε, τα ε, δικαιώματα των πολιτών και τα έχει καταδικάσει αυτά και το δικαστήριο. Και τώρα από την πίσω πόρτα ανοίγουμε κάποια δυνατότητα ή παραθυράκια. Είμαστε στεναρά αντίθετοι με οποιαδήποτε ε, απόπειρα να αποδυναμωθεί η προστασία που υπάρχει σήμερα. Έτσι κι αλλιώς οι τηλεπικοινωνίες διέπονται από το νέο καθεστώς και ρυθμίζονται. Και αν θέλετε να διαφυλάξετε οτιδήποτε αξίζει να συζητηθεί, ε, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι θα βελτιώνεται και δεν θα επιδεινώνεται η προστασία των πολιτών από τις υποκλοπές. Από την Ενωτική Αριστερά, η κυρία Κόνη Ένστ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι τούτη εδώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και χαίρομαι που την κάνουμε, αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει γιατί έπρεπε να αρχίσουμε από αυτό το θέμα. Αλλά ας αρχίσει έτσι η Προεδρία του Συμβουλίου. Θέλω να επανέλθω στην προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο. Γιατί έχει κολλήσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. ποια είναι τα προβλήματα. Θέλετε να το γιώσετε όλο αυτό και να προχωρήσετε σε κάτι άλλο. Θέλω περισσότερες προφορίες. Ε, να πω και κάτι άλλο επί της αρχής. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία στο ίντερνετ, να προχωρήσουμε σε ποινικά μέτρα, γι' αυτό χρειαζόμαστε δεδομένα και μεταδεδομένα ε, επί παντός επιστητού. Μιλάμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε μαζικά και συλλογικά. Όλο και περισσότερο μου λείπει το να λέμε με την ίδια ανάσα, με την ίδια ανάσα όμως για την προστασία των πολιτών και να μην το θεωρούμε κάτι ενοχλητικό ή κάτι σχετικό, ε, να αρχίσουμε να μιλάμε για αποκρυπτογράφηση κτλ. Ε, για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα μπορούσατε λίγο να μας το σχολιάσετε και αυτό υπάρχει μια δυσαναλογία ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων και μετά την υποτιθέμενη ανάγκη για τόσα πολλά δεδομένα που πρέπει και να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε. Αυξάνεται αυτή η ανισορροπία και ειδικά στο Συμβούλιο βλέπω και πολλές διαφωνίες με τη θέση του Κοινοβουλίου. Η παρακολούθηση πια έχει καταντήσει μαζική, χωρίς να υπάρχει παραμικρή υποψία. Έτσι γενικά ένα φακέλωμα. Έχουμε το γενικό κανονισμό, έχουμε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εσείς τι θα κάνετε για να επανέλθει αυτή η ισορροπία. Έχετε καμιά τέτοια πρόθεση. Για να υπάρχει κάποια σχέση λογική Εντάξει, καταλαβαίνω ότι στα ποινικά και στην τρομοκρατία χρειάζεται να συλλέγουμε κάποια δεδομένα. Δεν είμαστε εμεί αντίθετοι. Αλλά ε, υπάρχει προστασία των δεδομένων που καταργείται κάθε φορά με διάφορες προφάσεις. Εσείς που θέλετε να αφήσετε το στίγμα της Προεδρίας σας. Ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό να το Ευχαριστώ πολύ. Έχει στήσει το λόγο από το ΕΛΚ Ο κύριος Γκρέσλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριος Γκρέσλερ, Ευχαριστούμε και τον ε, Υφυπουργό για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κροατικής Προεδρίας και το ζήτημα αυτό. Έχω ένα ερώτημα να θέσω στα κροατικά. Γίνονται πολλές συζητήσεις σήμερα για την θέσπιση νέων κανόνων με βάση τον κανονισμό αυτό η privacy γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι μεγάλο μέρος της συζήτησης αυτής ε, έγινε και στα πλαίσια της εισαγωγής της νομοθεσίας GDPR. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιους κανόνες έτσι ώστε οι χρήστες ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών να μπορούν να χαίρουν τα υψηλότερα πρότυπα, τι πρώτε προδιαγραφές προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τη χρήση νέων τεχνολογιών, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους ε, ε, χρήσης, ε, κακής χρήσης των, ε, των μέσων αυτών, ιδιαίτερα για τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες, ε, τα παιδιά. Στην Κροατία, στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, έχει υποβληθεί μία πρόταση για την e-privacy και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε λύσεις. Το ερώτημά μου είναι ποια είναι συγκεκριμένα τα σχέδια για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τον φάκελο αυτόν και πότε σκοπεύετε να φτάσετε σε συμφωνία και με το Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή νομίζω 15 κράτη-μέλη είναι αντίθετοι με το παρόν κείμενο. Ναι, θα θέλαμε βεβαίω να πούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να πάρει το λόγο. Μάλιστα, κάποιο ε, αναφέρθηκε στην Κομισιόν και στι αρμοδιότητε τη ε, νωρίτερα. Θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. έχουμε κάποια σχόλια να κάνουμε σε σχέση με αυτά που συζητήθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τους στόχους της προστασίας ε, της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών, όλων των επικοινωνιών και όχι μόνο τα metadata, όλων των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, ε, η Κομισιόν, ε, είπαμε ότι η Κομισιόν δεν θα επικρίνει το Συμβούλιο εάν καθυστερήσει. εάν πραγματικά Υπόθηκε αυτό, αλλά ρωτήστε πόσες φορές έχουμε πει ε, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να τα βρουν, πρέπει να αρχίσει η διαπραγμάτευση η διαθεσμική. Το είπαμε στην Κορεπέρ, το είπαμε στις συνεδριάσεις ε, στο Συμβούλιο, στις Υπουργικέ Συνόδους, στις ομάδες εργασίας. Οπότε δεν νομίζω να ισχύει αυτό που ελέγχθη. Τώρα το ερώτημα του κατά πόσο η Κομισιόν εξετάζει το θέμα της εφαρμογής ή όχι. Εμείς ρωτήσαμε πέρυσι τα κράτη-μέλη πώς η εφαρμογή της οδηγίας, του κανονισμού της οδηγίας αυτής ε, είναι, είναι συμβατή με το GDPR. Και μια σειρά από άλλε ερωτήσει τη εφαρμογή αυτών των νομοθεσιών σε εθνικό επίπεδο. Έτσι. Χρειάζονται κάποιε διευκρινήσει. Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα και από με τα κράτη-μέλη, παρακολουθούμε την εφαρμογή των σχετικών νομοθετημάτων. Επίση, ε, ελέγχθη ότι η Κομισιόν θέλει να, υπάρξει, να, αποσυρθεί δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και από αυτά που έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι σαφές ότι για μας είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτού του φακέλου. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο κύριε Μπιλαβέρ για να απαντήσετε στα ερωτήματα και τα σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας και για τη συζήτηση, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι, γιατί περισσότερο είχαμε σχόλια παρά ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ όμως ε, για όλα και για την ε, συμμετοχή της Κομισιόν. Η συζήτηση σήμερα δείχνει ξεκάθαρα πόσο δύσκολος είναι ο φάκελος αυτός και πόσο δύσκολο θα είναι να βρούμε μία λύση. Όλες οι αμφιβολίες που κατατίθενται σήμερα δεν είναι εύκολο να επιληθούν. Ξέρουμε τώρα γιατί οι προηγούμενες 7 προεδρίες είχαν προβλήματα στο να καταλήξουν σε συμβαστική λύση. Όμως, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν θα πρέπει να αλληλοκταξεύουμε κατηγορίες γιατί όλοι είμαστε εδώ και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε όλοι ένα κοινό στόχο, την προστασία της ιδιωτικότητας. καθώς και την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Το να βρούμε μια φόρμουλα να το επιλύσουμε αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Θα έλεγα ότι είναι ένα είδος αλχημίας. Δεδομένου το ότι οι προηγούμενες 7 προεδρίες δεν κατόρθωσαν να βρουν την κατάλληλη φόρμουλα, θα ήταν κάπως αλαζονικό από την πλευρά μας να πούμε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Όμως, τι μπορώ να σας υποσχεθώ από την πλευρά της Προεδρίας, ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας θα λάβουμε υπόψη και τη σημερινή συζήτηση και όλα τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί. Θα λάβουμε υπόψη και τη συζήτηση που είχαμε στο Συμβούλιο το Δεκέμβριο, όπου ακούσαμε τα 15 κρατημέλη γιατί συμφωνούν με ορισμένε διατάξεις. Και κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου θα προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικότητας και της ανάγκης για καινοτομία και για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Το Φεβρουάριο λοιπόν θα παρουσιάσουμε το νέα συμβαστική μας πρόταση και αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι σε διάλογο με όλα τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και να βγούμε από το τέλμα και να πετύχουμε πρόοδο. Κάτι στο οποίο απέτυχαν οι άλλες προεδρίες στο παρελθόν. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, για τις ερωτήσεις. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα με συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ και πραγματικά ευχόμαστε αυτό το εξάμεινο να μπορέσει να σημάνει πραγματικά την απεμπλοκή σε αυτό το σημαντικό φάκελο σας. Ευχαριστούμε κύριε Υφυπουργέ και ευχαριστούμε και την ομάδα σας. Να περιμένουμε πέντε λεπτά πριν να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Μπορείτε να ξεκουραστείτε για λίγο. Bien, Eh, queridos colegas, vamos a... Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο 13ο σημείο της ημερησής διάταξης που έχει να κάνει με τα τεχνικά και δικαστικά προβλήματα με τα δεδομένα τηλεπικοινωνιών στη Δανία και τη χρήση εσφαλμένων ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικέ καταδίκες. Όπως ε, γνωρίζετε, οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο του 2019, σύμφωνα με τις οποίες οι δανεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 10.700 ε, καταδίκες ε, ποινικών δικαστηρίων από το 2012 θα αναθεωρηθούν λόγω σφαλμάτων ε, στα συστήματα τηλεπικοινωνιών. Ε, είναι πραγματικά μια ανατριχιαστική είδηση. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 η εστάλη στην ε, Κομισιόν μια κοινοβουλευτική ερώτηση ε 00267319 που δεν φαίνεται να έχει λάβει ακόμη απάντηση. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τον ε, επικεφαλής ε, ε, της προστασίας ιδιωτικής ζωής και δεδομένων της εθνικής αστυνομίας και τον Διευθυντή Ένωση Τεχνολογία Πληροφοριών και Πολιτική Ζωνίας. Σα ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση τη Επιτροπή αυτή. Για... Τη Επιτροπή Ελευθεριών Δικαιοσύνης στον Κοινοβουλίο καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάσπερ Λούν, ο οποίο είναι διευθυντή τη Ένωση Τεχνολογία και Πληροφοριών και Πολιτική τη Δανία, για να μα δώσει κάποιε εξηγήσει σχέση με την υπόθεση. Έχετε το πολύ 10 λεπτά, κύριε Λούντ, αν έτσι προφέρετε το όνομά σα, σα ευχαριστώ για την παρουσία σα εδώ και έχετε το λόγο. <clears throat> Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ευθεριών, σας ευχαριστούμε που με καλέσατε να μιλήσω για την υπόθεση αυτή της ε, Μονάδας Προστασίας Δεδομένων. Ε, υπάρχει μια οργάνωση κοινωνίας των πολιτών η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό, την ειδική μας. Είμαστε μέρος ε, και της σχετικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά από τις αρχές επιβολής δεδομένων ε, επιβολή του νόμου, συγγνώμη, είναι ε, βασικό ζήτημα που μα απασχολεί από τα, την αρχή του 2000. Αυτά τα δεδομένα μας οδηγούν σε πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα για κάποια άτομα, τις σχέσεις που έχουν, το που διαμένουν και βεβαίως ε, το πώς μετακινούνται και προ τα που μετακινούνται. Η πρόσβαση στα στοιχεία τηλεπικοινωνία από τι αρχέ επιβολή του νόμου βεβαίω δημιουργεί ανησυχίε ε, για τα αισθήματα ιδιωτικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων και αυτό αναγνωρίζεται και στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μια σοβαρή ανησυχία σχετίζεται με το γεγονό ότι τα δεδομένα του επικοινωνίου χρησιμοποιούνται από τι αρχέ επιβολή του νόμου. Ε, μπορεί να μην είναι σωστά λόγω λαθών που υπάρχουν από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών οι αρχέ επιβολή του νόμου, λοιπόν, ορισμένε φορέ μπορεί να φτάσουν σε λάθο συμπέρασματα λόγω των δεδομένων αυτών και να θεωρούν ότι το προφίλ ε, τη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών είναι ακριβή. Είναι, είναι ακριβέ. Και έτσι μπορεί ε, κάποιοι άνθρωποι να διώκονται ε, ενώ είναι αθώοι. Αυτέ οι πτυχέ τη χρήση των δεδομένων των επικοινωνιών από τι αρχέ επιβολή του νόμου δεν εξετάζεται επαρκώ στην υπάρχουσα συζήτηση υπάρχει μια τάση να θεωρούμε ότι τα στοιχεία από την επικοινωνίες είναι σωστά ε, διότι προέρχονται από μηχανήματα, δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση. Το σενάριο όμως με τα λάθος δεδομένα συνέβη σε μαζική κλίμακα στην Δανία πριν από μερικά χρόνια. Το πρόβλημα με τα λάθος δεδομένα ε, το ανακαλύψαμε το 2018, αλλά ε, το αποκαλύψαμε στο, ευρύ κοινό τον Ιούνιο 2019 υπήρξε μια εσωτερική έρευνα στο επίπεδο αστυνομία και σιγά σιγά ε, καταλάβαμε το μέγεθο του προβλήματο. Τον Ιούλιο του 2019 φτάσαμε στο συμπέρασμα από ότι από τι 8.500, περίπου 8.500 έρευνε είχαν επηρεαστεί από αυτά τα λανθασμένα δεδομένα από το 2012. Ο αριθμός 12.000, συγγνώμη, 12.700 περιπτώσεις ε, είναι αυτέ ε, όπου ξέρουμε σίγουρα ότι ε, στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν στι ιδιωτικέ έρευνε. Δεν σημαίνει, είναι ο αριθμό των ατόμων που στη συνέχεια βέβαια υπέστησαν διώξει. Ε, το Σεπτέμβριο του 2019 ε, είχαμε πρώτα ένα μορατόριο για δύο μήνε στη χρήση των δεδομένων τηλεπικοινωνιών στι ποινικέ δίκε και στην προδικαστική διαδικασία. Αυτό το δραστικό μέτρο για τη μη χρήση στοιχείων τηλεπικοινωνιών ε, έπρεπε να πάρθει. Η βασική πηγή πληροφοριών για το τι συνέβη είναι μια έκθεση από την Deloitte που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και που ζητήθηκε από τη Δανική Αστυνομία τέλη Αυγούστου. Για να είμαι σύντομος, τα λάθη σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών είχαν να κάνουν με τη Δανική Αστυνομία αφότου ελάμβαναν δηλαδή τα στοιχεία από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Έδιναν τα στοιχεία οι παροχοί σε διάφορες, σε διάφορες τεχνικές μορφές και η ιδανική ε, αστυνομία τα, τα μετέτρεπε σε ένα συγκεκριμένο format και υπήρχε ένας timer, ένας χρονοδιακόπτης ε, που ε, χρησιμοποιούσε ο αστυνομικό εξωματικό πριν ολοκληρωθεί η μετατροπή ορισμένε φορέ. Και αυτό οδηγούσε σε ελλειπή δεδομένα, έλειπαν στοιχεία δηλαδή από αυτά που προερχόντουσαν αρχικά από του παρόχου. Ήταν άλλε οι συνισταμένε οι γεωγραφικέ επίση από, το σύστημα, από ένα σύστημα στο άλλο και αυτό οδηγούσε σε περαιτέρω λάθη. Όπω περιέγραψα, είναι εύκολο να διορθωθούν τα λάθη αυτά. Αρκούσε δηλαδή να ε, από ε, αποσυνδεθεί ο χρονοδιακόπτης αυτός. Είναι όμως περίπλοκο το σύστημα αυτό, είναι ξεπερασμένο. Τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των επικοινωνιών αυτών είχαν αναπτυχθεί από την, εθνική αστυνομία της Δανίας από έναν και μόνο υπάλληλο σε εσωτερικό επίπεδο χωρίς διαβούλευση. Ε, πριν τον Δεκέμβριο του 2019 δεν υπήρχε καμιά διοικητική πρακτική σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτή τη μετατροπή των δεδομένων. Από κοινού την έκθεση του Deloitte, το Υπουργείο Δικαιοσύνη ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Δύο εβδομάδε αργότερα σταμάτησε αυτό το moratorium. Επανήλθαμε λοιπόν ε, στην κανονικότητα. Ε, Μπορεί να χρησιμοποιηθούν πλέον τα στοιχεία αυτά από την Δανική Αστυνομία και στι δίκε. Βεβαίω ε, τα προβλήματα, τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την ξεπερασμένη, ξεπερασμένη υποδομή πληροφορική. Θα χρειαστεί χρόνο για να αναπτύξουμε νέα πληροφορικά συστήματα. Θα γίνουν μια σειρά από ελέγχου βέβαια από ανθρώπινο χέρι αυτή τη φορά. Όμω ε, θα πρέπει να δούμε πώ θα χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα στι αστυνομικέ έρευνε στο μέλλον. Τώρα μια σειρά από νομικούς, δικαστές, δικηγόρους θα ενημερωθούν ε, από την Deloitte για τη χρήση των δεδομένων σε ποινικέ υποθέσεις. Αυτή η ενημέρωση θα εξετάσει, θα εξηγήσει τη βασική χρήση των δεδομένων αυτών από τις αστυνομικές αρχές και πληροφορίες για το πώς τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τα δίκτυα τηλεφωνικής ε, ε τηλεφωνίας. Αυτό είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, τα, οι κινητές συσκευές δεν συνδέονται απαραίτητα με κάποιο ε, tower Δηλαδή μπορούμε να θεωρούμε ότι κάποιος είναι κοντά ε, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία με βάση τα δεδομένα, αλλά δεν είναι ακριβές αυτό. Δεν είναι απαραίτητα κοντά στην κεραία δηλαδή. Και ορισμένες φορές ε, και οι αστυνομικοί αλλά και οι εισαγγελείς ε, υπερβάλλουν στο, στην εμπιστοσύνη που δίνουν στην ακρίβεια αυτών των γεωγραφικών δεδομένων. Υπάρχει μια task force αυτή τη στιγμή που προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει Αυτέ τι 12.000 ε, περιπτώσει που ενδεχομένω να έχουν επηρεαστεί από αυτά τα λάθη ε, των στοιχείων αυτών. Μια ανεξάρτητη διευθύνουσα ομάδα υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνη θα παρακολουθεί αυτή την task force. Ε, το έργο αυτό, οι εργασίε αυτέ είναι εξελίξη. Δεν μπορώ να πω κάτι δηλαδή για αυτά. Θα πρέπει όμω να δούμε τελικά πώ χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα στοιχεία τηλεπικοινωνία στην κάθε υπόθεση και πώ αυτό ε, βεβαίως θα περιπλέξει το έργο τη Task Force το να μπορούμε να τα υπεριθέψουμε όλα αυτά ενώ ε, τι μάθαμε λοιπόν από, αυτήν, από αυτό το σκάνδαλο με τα στοιχεία τηλεπικοινωνιών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στον κίνδυνο λάθου στα στοιχεία τηλεπικοινωνιών όταν το, το, τα χρησιμοποιούν οι αρχέ που στον νόμο Αυτό ισχύει για όλου. Ε, Στι αρχιδιοπτικέ αρχέ, εισαγγελεί, δικαστέ, δικηγόροι. Επίση είναι σημαντικό και για τη συζήτηση το ποια είναι τα, τα δεδομένα αυτά που μπορεί να, να παρακρατούμε και ποια όχι ε, και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. νομίζω ότι η εμπειρία που έχουμε μετά από αυτή τα συστημικά, συστηματικά λάθη ε, να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να μην ε, παραλευθούν τέτοια πράγματα είτε στην Δανία είτε αλλού. Υπάρχουν όμως και άλλες πηγές λαθών ή κακής ερμηνείας ε, στοιχείων από αρχέ επιβολή του νόμου, τα το, οποία, προέκυψαν στην περίπτωση τη Δανία. Πρέπει πάντα να τονίζουμε ότι τα δεδομένα ε, έχουν να κάνουν με μια υπηρεσία τηλεπικοινωνίας. Η, η, χρήση αυτών των δεδομένων από αστυνομικές αρχές είναι μια δευτερογενής πλέον, ένας δευτερογενής στόχος ε, η μορφή χρήσης και δεν είχα προβλεφθεί γι' αυτό τα δεδομένα αυτά. Και θα, θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει στο ότι τα δεδομένα θα δίνετε λιγότερη σημασία σε κάποια προσωπικά δεδομένα. Επίσης, υπάρχουν νέε τεχνολογίες κινητής ε, ε και τηλεφωνίας, ε, LTE, το, σε ό,τι αφορά το Wi-Fi επίσης. Και εκεί μπορεί να οδηγηθούμε σε λάθη εφόσον δεν υπάρχει σαφή αναγνώριση κατά τη δευτερογενή αυτή χρήση όταν τα ίδια αυτά στοιχεία τα επεξεργάζονται δηλαδή οι αρχές επιβολής του νόμου. Ολοκλήρωσα με την εισαγωγή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Sí, muchísimas gracias. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κρίστεν Ισχάμπερ από την αντίστοιχη μονάδα της Εθνικής Αστυνομίας της Δανίας. Έχετε το λόγο για να μας ενημερώσετε για τα μέτρα που λάβατε ή που πρόκειται να λάβετε για να λυθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία έχετε εντοπίσει και σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω την Επιτροπή σας για αυτά τα συμβάντα ε, στη Δανία ως προς τα δεδομένα. Πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα με πολύ μεγάλη σοβαρότητα ε, από πλευρά της αστυνομίας, λέει ο κύριος Βίσες Φάνμπεργκ. Πρόκειται για ποινικέ υποθέσεις που βρίσκονται στη δανική δικαιοσύνη αυτό τον καιρό και φυσικά ε, εμείς έχουμε την ευθύνη να μην προσάγονται στη δικαιοσύνη και να μην καταδικάζονται αθώοι η αστυνομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί ε, σωστά αποδεικτικά στοιχεία και γνήσια. Υπάρχει φυσικά και το τεκμήριο της αθωότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγιναν λάθη στη μετατροπή των δεδομένων, στη μεταφορά τους από τις τηλεκοινωνίες και τότε τι να κάνουμε, δεν ήταν αρκετά ε, καλός ο έλεγχος ποιότητας, ούτε η τεκμηρίωση, ούτε οι αποδείξεις, ούτε καν οι για πιθανά σφάλματα. Συστηματικά είχαμε υπό εκπροσώπηση, ε, κανένας δεν καταλάβαινε ότι ήταν λάθη αυτά που γινόντουσαν ε, και είχαμε κάποιους παρόχους τηλεπικοινωνίας που ε, υπόκεινται ένα ένα πλημελή έλεγχο πολλά χρόνια και όλο και περισσότερο σε ποινικέ υποθέσεις χρησιμοποιήθηκαν ε, στοιχεία από την τηλεπικοινωνία που κανένας δεν είχε αναγνωρίσει ότι ήταν ε, πλαστά ή ότι δεν ήταν ε, ορθά. Ούτε οι εισαγγελεί, ούτε οι συνήγοροι, ούτε κανένας. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα και πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να ανοιχνευθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία ω προ την επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων από την αστυνομία. Υπάρχουν ε, συνάδελφοι που είναι πάρα πολύ ειδικοί και πεπειραμένοι σε αυτά. Ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ποιο ήταν το πλαίσιο και πώς ε, ε, δίδονται, διαβιβάζονται αυτά τα στοιχεία. Σύμφωνα με τον νόμο στη Δανία ε, μπορεί η αστυνομία μετά από δικαστική παραγγελία να παίρνει στοιχεία από εταιρείε κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει άρση απορρίτου και μπορείς να δεις ποιος έχει τηλεφωνήσει σε ποιον ένα κινητό που βρισκόταν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από κάποια κέντρα λοιπόν τηλεπικοινωνιών η αστυνομία ζητάει αυτά τα στοιχεία, τα στέλνουν οι εταιρείε ε, κινητής τηλεφωνίας εφόσον τα έχουν ε, και παίρνουν κάποια στοιχεία από το διαδίκτυο ε, και μας τα δίνουν υπό μορφή hidden, bulk data από αυτά Δηλαδή δεν πρέπει ο πάροχος να δίνει στην αστυνομία σε ένα συγκεκριμένο format αυτά τα στοιχεία, μας τα στέλνουν έτσι σόριδον και από εκεί και πέρα η αστυνομία επιφερτίζεται με το έργο να τα ε, αξιοποιεί, να τα μετατρέπει για τις διάφορες ποινικέ υποθέσεις. Δηλαδή ε, τα λαμβάνουμε με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο, format, μορφότυπο, ε, υπάρχει ένας αριθμός σειρών στοιχείων και ε, ε, για κάποια δραστηριότητα ε, σε κάποια δραστηριότητα αντιστοιχεί ένας αριθμός σειρών. Πρέπει να αλλάξει το format και αντιστοιχεί πάντα αυτό σε μία κεραία που έχει πιάσει το σήμα ενός SMS. Αυτά τα στοιχεία τα δίνουν στην αστυνομία, τα διαβιβάζουν Και έχουμε δύο σετ, ας πούμε, δεδομένων. Τα, ε, τα μεν είναι αυτά που παίρνουμε σε μορφή ε, χωρίς επεξεργασία και η δεύτερη είναι επεξεργασμένη μορφή. Την, την 1η Δεκεμβρίου 2010, λοιπόν, αυτό το τηλεφωνικό κέντρο διαβίβασε τα στοιχεία στην αστυνομία. Και όπως σας είπα, κανονικά Υπάρχει ένας αριθμός σειρών που αντιστοιχεί σε κάποια στοιχεία και τα αντιπαραθέτουμε για να δούμε ποια μας, δεδομένα μας έχουν ε, μεταδώσει. Εκεί λοιπόν επανειλημμένα είδαμε ότι δεν συμφωνούσαν τα χείριν στοιχεία με τα ε, στοιχεία που είχαν προκύψει από τη μετατροπή, ο αριθμός των σειρών, σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εδώ υπάρχουν τρία σενάρια. Ε, ε, ίσως δεν ήταν η σωστή ε, παροχή όλων των στοιχείων και υπάρχει λάθος στο σύστημα τηλεπικοινωνιών ή υπάρχει λάθος στο σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων είτε η ανάλυση ήταν λάθος και ήταν λάθος η μετάδοση των στοιχείων. Το πρώτο λάθος που διαπιστώθηκε το 2019 ήταν λάθος του συστήματος τηλεπικοινωνιών και μάλιστα συστηματικά Γι' αυτό είχαμε και διαφορές ανάμεσα ε, ε, στα στοιχεία που παίρναμε που ήταν ακατέργαστα ας πούμε και στα κατεργασμένα στη συνέχεια. Και το σύστημα αυτό ε, ευθύνεται για τα λάθη. Είπαμε ότι υπήρχε ένας χρονοδιακόπτης, τα ημέρα ακούσαμε, στο σύστημα αυτό της τηλεπικοινωνίας και κατά τη λήψη και κατά την επεξεργασία. Υπάρχει ένα timer ε, το οποίο ε, εισήχθη στο σύστημα για να μπορούν να μεταδίδονται αυτά τα στοιχεία ε, και τα δεδομένα στα διάφορα αστυνομικά τμήματα. Και θα πρέπει ε, το συντομότερο, αυτό ήταν ο στόχος μας, ε, να μεταδίδονται αυτά τα δεδομένα στην αστυνομία, στα διάφορα επιμέρους αστυνομικά τμήματα. Αυτό ήταν το λάθος, τη μετατροπή. Ε, δηλαδή, ακούσατε ότι ο διακόπτης σταματούσε ε, τεχνητά ε, πριν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των δεδομένων για να μεταδοθούν ε, σε ένα αστυνομικό τμήμα, οπότε ήταν λάθος τα στοιχεία, γιατί δεν περίμεναν να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Αυτή ήταν μία πηγή λάθος. Υπήρχαν και άλλες όμως ότι δεν ήταν πλήρη αυτά τα δεδομένα. Αυτό το πρόβλημα το αναγνώρισαν, κατάλαβαν ότι είναι ο χρονοδιακόπτης και ε, τον έκλεισαν, σταμάτησαν τη λειτουργία του. Τώρα για τις μεμονωμένες ποινικέ αυτές οι υποθέσεις. Ε, καταλάβαμε ότι υπάρχει αυτό το σφάλμα, το εντοπίσαμε και στις 13 Ιουλίου του 2019 αποφασίσαμε να ξαναδούμε όλες αυτές τις ποινικέ υποθέσεις όπου ενδεχομένως να είχε παρισφρήσει αυτό το λάθος και να είχε συνέπειες πάνω από 10.000 υποθέσεις από την 1η Πρώτου του 2012 μέχρι τις 18 Τρίτου 2019. Εξετάσαμε ξανά όλες αυτές τις υποθέσεις. Φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί γίνεται και με το χέρι αυτό, δεν είναι αυτόματο. Θα ακολουθήσει ΕΔΕ, έρευνα και έκθεση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι σε προσωρινή κράτηση προφυλάκηση ε, ή που ε, ε, μπορούν να κάνουν καταγγελίες. Οι ορισμένοι έχουν ήδη δικαστεί, έχουν καταδικαστεί. Φυσικά αυτά είναι ύψιστη προτεραιότητα για όσους έχουν ήδη καταδικαστεί. Δεν έχουμε εντοπίσει ε, κάποιο τέτοιο σφάλμα όπου ε, ακριβώς λόγω αυτού του λάθους στα δεδομένα και στις τηλεπικοινωνίες να ε, οδηγηθήκαμε σε δικαστική πλάνη και να καταδικάστηκε κάποιος αθώος. Στις 2 Ιουλίου 2019 συστάθηκε μία ανεξάρτητη ομάδα ελέγχου και συντονισμού για να εξετάσουν αρμοδίως την κατάσταση και να, να ελέγξουν τις αρμόδιες αρχές και να υπάρχει και πλήρης πρόσβαση του κοινού, να είναι δημόσιο αυτό και να έχουμε και στοιχεία εξωτερικού ελέγχου ε, για τη λειτουργία και τη συμπεριφορά των διοκτικών αρχών. Πρόεδρος εκεί είναι ένας δικαστής, μετά συμμετέχουν δύο συνήγοροι, δικηγόροι περάσπισης, ε, ε, κάποιος που είναι ειδικό για τις αστυνομικέ έρευνες και καθηγητές νομικής. Επίσης έχουν και εξωτερική υποστήριξη από ειδικού ηλεκτρονικών υπολογιστών στις 18 Αυγούστου. Δόθηκε μια εντολή για την πρόσβαση σε δεδομένα ε, διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Ε, μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Επίσης, τον Αύγουστο 2019 ανατέθηκε μια εξωτερική μελέτη για να εντοπίσουμε το συντομότερο ε, την πηγή του σφάλματος, για να μπορούν να εξαχθούν τα αντίστοιχα συμπεράσματα και να μπορούμε να τρέχουμε ξανά στις ποινικέ υποθέσεις σε τέτοια μεταφορά δεδομένων και επεξεργασία. αφού έγιναν όλα αυτά, επετράπη και πάλι η χρήση με τη νέα μορφή αυτής της διαδικασίας και ε, ορίζεται σαφώς τι μπορούν να κάνουν οι πολιτικοί, οι εισαγγελίες, η αστυνομία, οι δικηγόροι, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικέ υποθέσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία από τις τηλεπικοινωνίες και τα δεδομένα που αφορούν πολίτες. Και τον Οκτώβριο του 2019 το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες ε, και εξέδωσε συστάσεις και εντολές για να μπορούμε και πάλι να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους δεδομένα ως αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχει και πλήρης περιγραφή, αν σας ενδιαφέρει, της κατάστασης. Ε, επίκειται νομοθετική πρόταση, ακριβώς για να μπει και ένα στοιχείο υποχρεωτικής επίβλεψης και ελέγχου. για να εξοπλιστεί καλύτερα το κέντρο δεδομένων της αστυνομίας με περισσότερα μέσα, με πιο επαγγελματική λειτουργία και υποστήριξη για να γίνεται και ο αντίστοιχο ποιοτικό έλεγχος. Το κέντρο επεξεργασίας δεδομένων δηλαδή, για να μην επαναληφθούν τέτοια σφάλματα. και για κατάρτιση, επόκτηση δεξιοτήτων για τις διοκτικές αρχές και την εισαγγελία. Αυτό το συμφωνούν και με τις αρμόδιες ενώσεις δικαστικών, ε, το Δικηγορικό Σύλλογο κλπ. Έχουν ήδη ληφθεί κάποια μέτρα και πρέπει να το τονίσω. Βέβαια αυτό ήταν σκάνδαλο και έχει γίνει μεγάλος άλλος για το πώς και κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται τέτοια δεδομένα σε ποινικέ υποθέσεις ως αποδεικτικά στοιχεία. Και έχουν προσθεθεί και νέες πρωτοβουλίες. Αυτά, αν έχετε ερωτήσει με χαρά να απαντήσω αν μπορώ. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται. Και αν θέλετε και περισσότερες λεπτομέρειες στη διάθεσή σας. Bien, le agradecemos también a σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Γενική Διευθυνσή. Home έχει το λόγο κύριος Λόταρς. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν γνωρίζει το θέμα αυτό από τότε που δημοσιεύθηκε πριν στο καλοκαίρι. Η πρώτη μας κατανόηση με το πρόβλημα στην Δανία ήταν ένα πρόβλημα τεχνολογίας των πληροφοριών με το σύστημα που μετατρέπει τα δεδομένα ε, σε αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, σε δικαστικές ε, υποθέσεις. Παρακολουθήσαμε λοιπόν στενά την υπόθεση και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Αργότερα συνειδητοποίησαμε όταν δημοσιεύτηκε και η εξωτερική έκθεση της Deloitte ότι ένα άλλο ζήτημα ήταν η έλλειψη της κατάλληλης αξιολόγησης ή των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας. Η κατανόηση της Κομισιόν, επομένως, είναι ότι είναι τεχνικά ή οργανωτικά διαδικαστικά τα θέματα στην ε, αστυνομία της Δανίας και στο δικαστικό σύστημα και δεν προκύπτουν από ελαττώματα ή ελλείψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, ή των ε, ηλεκτρονικών αποδεκτικών στοιχείων. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ε, την σημασία του θέματος αυτού και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η ποιότητα της, και το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων στις ε, εθνικές δικαστικές διαδικασίες ε, καλύπτονται από εθνική νομοθεσία και τα θέματα που έχουν να κάνουν με το παραδεκτό των αποδεκτικών στοιχείων ε, ή της επαρκούς ή μη επαρκούς ποιότητας θα πρέπει να αξιολογείται από τα εθνικά δικαστήρια. Εμείς επομένως ως Κομισιόν δεν είμαστε αρμόδιοι να αξιολογήσουμε το θέμα αυτό να αξιολογήσουμε την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων και τη ε, χρήση των ε, δεδομένων αυτών ε, στις δικαστικές διαδικασίες. Αυτό πρέπει να γίνει από τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια. Αυτό που θέλουμε όμως να σημειώσουμε σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι ο νόμος, ο Ευρωπαϊκός Νόμος Προστασίας των Δεδομένων και στη συγκεκριμένη κατάσταση ή οδηγία για την προστασία των δεδομένων ε, σε σχέση με την επιβολή του νόμου καθιστά σαφές ότι η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτή η αρχή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ένα πλαίσιο επιβουλής του νόμου και σε ένα δικαστικό πλαίσιο. Και φυσικά αναγνωρίζεται αυτό από την Κομισιόν. Αυτή η αρχή θα πρέπει να ισχύει Επίσης, ε, η παρακολούθηση και η ποιότητα των δεδομένων εγγράφονται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και εμείς ως Κομισιόν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά δεν είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση επί του συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή δεν έχουμε αρμοδιότητα να εξετάσουμε θέματα ποιότητας δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς ε, δεν έχετε αρμοδιότητα να εξετάσετε την ποιότητα των δεδομένων. Όμως ε, η Κομισιόν μπροστά σε μια τέτοια υπόθεση κάτι θα μπορούσε να φανταστεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι κάτι τόσο σοβαρό σε μια προηγμένη χώρα όπως η Δανία θα πρέπει να τραβήξει την προσοχή μας ως κάτι έκτακτο, κάτι εξαιρετικό και ίσως ε, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Θα δώσω το λόγο στη συντονίστρια του Ρινιού που είναι εδώ παρούσα και κατόπιν ε, στους βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Ίντβελτ. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μιλάω και ως ε, συντάκτρια της ε, ερώτησης προς την Κομισιόν που δεν απαντήθηκε. Μάλλον θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να ασχολείται με τις ερωτήσεις που υπογράφει η κυρία Ίντφελτ, γιατί ποτέ δεν λαμβάνω απάντηση. Και μετά έρχεται η Κομισιόν εδώ και τελικά δεν με καθησυχάζει, με κάνει να ανησυχώ ακόμη περισσότερο. Θα επανέλθω στην ίδια την κοινοβουλευτική ερώτηση σε ένα λεπτό. Και φυσικά θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν γιατί δεν απάντησε. Ανησυχώ πάρα πολύ από την απάντησή σας. Αν σας ακούω να λέτε «Α, μια χαρά ήταν η νομοθεσία», το πρόβλημα ήταν στην εφαρμογή. Τότε η νομοθεσία δεν είναι καλή γιατί δεν υπάρχουν απαραίτητε ασφαλιστικέ δικλείδε. Γιατί αν ήταν επαρκείς οι ασφαλιστικές δικλείδες, τότε δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί αυτό. Επίσης, νομίζω να στην οδηγία περιδιεκτικών ερχών που αφορά την προστασία των δεδομένων, αλλά θέλω να τονίσω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν εφαρμόζουν την οδηγία αυτή, αλλά αντίθετα εργάζονται με την απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων που χρονολογείται από το 8. Τότε δεν υπήρχαν καν τα έξυπνα τηλέφωνα. Αλλά αυτό που στην πραγματικότητα με ανησυχεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, ουσιαστικά αναγάγει σε θρησκεία την διατηρήση των δεδομένων ε, γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να διευνήσει μία νέα δυνατότητα να προτείνει μια νέα οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων αφού οι προηγούμενοι για πολύ καλούς λόγους ε, ήταν αντικείμενο έντονης κριτικής από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλει η Κομισιόν λοιπόν να προτείνει μια καινούρια και κάνει μια ανάλυση για να προετοιμάσει την ελόγηση για μια νέα νομοθετική πρόταση. Και αυτό είναι ο τρόπος που το κάνετε. Υποτίθεται ότι πρέπει να εμπιστεύουμε τον τρόπο δράσης της Κομισιόν στο θέμα αυτό. Δεν είναι σοβαρή αυτή η στάση. Και όπως είπε και η Πρόεδρος, ε, η Δανία σίγουρα δεν είναι μπανανία. Είναι μία από τις πιο προηγουμένες χώρες στον κόσμο. Και ξέρετε, μπορούν κάποια πράγματα να πάνε λάθος παντού. Αλλά θα έπρεπε αυτό να έχει προβλεφθεί στην νομοθεσία και να είναι τυφλή η Κομισιόν απέναντι σε τέτοιου κινδύνου. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτά που θα προτείνετε. Τώρα, για να επανέλθω σε συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά τη Δανία. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο κυρίους για την παρουσία τους εδώ και που είναι πρόθυμοι να απαντήσουν ερωτήσεις. Δεν ε, είμαι σίγουρη όμως ότι κατάλαβα καλά. Ίσως ε, είπατε ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις ή παθέσεις όπου θα κατέληγε το δικαστήριο σε άλλα συμπεράσματα, γιατί αν κατάλαβα 32 άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί μετά από τις ανακαλύψεις αυτές. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να ήταν ε, στη φυλακή και να ήταν αθώος, αλλά τι γίνεται με κάποιους ε, που δεν τους συλλάβαμε, κάποιους εγκληματίες που δεν μπορέσαμε να τους ανακαλύψουμε. μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Επομένω, συνεχίζετε να εργάζεστε με το θέμα τη διατήρηση τη αποθηκεύση των δεδομένων, αλλά μα είπατε ότι προσπαθείτε να λύσετε τα διάφορα προβλήματα που υπήρξαν. Σκεφτήκατε εντωμεταξύ να εργαστείτε με ίσως πιο καινοτόμα μέσα όπως ε, το Clearview παραδείγματο χάρη, το οποίο επίσης δοκιμάζεται και έχουμε τη χρήση της αναγνώρισης των χαρακτηριστικών ε, του προσώπου. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία, γιατί δεν πίσω από αυτό είναι η ίδια και ακούω ότι οι διοκτικές αρχές στην Ευρώπη το χρησιμοποιούν. Θα ήθελα να επανέλθω στην Κομισιόν και στην ερώτηση που θέσαμε. Η πρώτη ερώτηση ήταν, θα συμπεριλάβετε αυτά τα απορίσματα στην ανάλυση σας Αφού άκουσα τη δηλωσή σας, ανησυχώ σχετικά. Δεύτερη ερώτηση. Τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Τέλεμα Σύλληψη, ε, το σύστημα ε, για τα πενικά μητρώα, την ε, Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα. Ποια θα είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων αυτών. Τι αν ανταλλάσσονται αυτά τα δεδομένα και τα λάθη ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Είναι δύσκολο πραγματικά να διορθωθεί η κατάσταση. Πώς το βλέπει αυτό η Κομισιόν. Και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών, την αμοιβαία νομική συνδρομή και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία με τις τρίτες χώρες, με μη ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή που χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα διατήρησης των δεδομένων ανησυχούμε για όλα αυτά. Όχι επειδή λέμε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουν στην νομή να κάνει τη δουλειά τη, αλλά η ιδέα είναι να συλλάβουμε του εγκληματίε και να του καταδικάσουμε και όχι αθώου ανθρώπου. Και φυσικά και αυτά τα δύο είναι σε κίνδυνο. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τι απαντήσει σα. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κυρία Ιντερφελτ. Μόλι και ο πρόεδρο ε, τη Επιτροπή ε, να θέσω όμως και εγώ το ερώτημά μου. Δεν γνωρίζω εάν στην χώρα σας η υπόθεση αυτή ε, έφτασε στο Συμβούλιο και αν προλέπει η Κομισιόν το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά της Deloitte, της Deloitte και αυτά που ε, και εσείς μπορέσατε να διαπιστώσετε ως ε, απαραίτητες πρακτικές έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι δεν θα μπορέσει ε, μια τέτοια, ε, ένα τέτοιο μαζικό λάθος να μολύνει αν θέλετε δεκάδες, εκατοντάδες υποθέσεις που, που είναι στα δικαστήρια είναι θέμα κοινή λογικής αυτό που σας λέω οι νομοθέτες η εκλεστική εξουσία πρέπει πάντα να έχουν κατά νου αυτά που λέει η κοινή λογική, ο κοινό νους. Επίσης, η αλυσίδα ε, των διαφόρων απολυτικών στοιχείων είναι εξαιρετικά σημαντική σε μια υπόθεση. Όταν υπάρχουν σημαντικές παραβιάσεις εδώ, υπάρχουν, προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Ε, ορισμένες φορές υπάρχουν αποφάσεις ε, προφυλάκησης ε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους, να, να τους ε, επιβλήθηκαν ποινές λαθασμένα και υπάρχει το θέμα της ατιμορρησίας. Σε αυτές τις 12.000 υποθέσεις μιλάμε για υποθέσεις εξελίγματος χρήματος, δολοφονιών, ανθρωποκτονιών, σοβαρές υποθέσεις και σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές υπάρχουν περιπτώσεις όπου δικηγόροι θα μπορέσουν να πετύχουν την ακύρωση αποφάσεων, δεκάδων, εκατοντάδων περιπτώσεων, σοβαρών. Γιατί, διότι είναι, ε, είναι ε, ε, σημαντικά εγκλήματα όπως το χρήματο, χρήματος, διαφθορά κτλ θα μπορούσαν κάποιοι να θωωθούν λόγω διαδικαστικών ζητημάτων, δηλαδή εδώ. Και να δώσω το λόγο και στον πρόεδρο που είναι εδώ. Thank you. Dear colleague. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Μάιτε που προείδρευσε σε αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης και που μας βοήθησες να καλωσορίσω εδώ και τους ομιλητές Ο κύριος Μπράιερ έχει το λόγο αν δεν κάνω λάθος, παρακαλώ Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τους ομιλητές που ήρθαν εδώ να συζητήσουν μαζί μας και το... ποια είναι τα διδάγματα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό το σκάνδαλο των επικοινωνιών στην Δανία. 30 άνθρωποι απολευθερώθηκαν, έτσι, έτσι, από τη φυλακή. Αποφυλακίστηκαν. Είναι τεράστιο σκάνδαλο. Πρέπει να το εξετάσουμε και είναι κρίμα που δεν είναι εδώ η Προεδρία του Συμβουλίου, διότι και με αυτούς πρέπει να το συζητήσουμε. Εάν δούμε, όταν βλέπουμε τα ευρήματα της Επιτροπής σας, υπάρχουν κάποια πολύ ανησυχητικά πράγματα εδώ συστήματα ε, πληροφορικής τα οποία είναι ξεπερασμένα, τα οποία ε, είναι δύσκολο να τα συντηρήσει κανείς, τα συντηρεί ένας και τα εξεργάζεται μόνο ένας άνθρωπος στο αστυνομικό τμήμα, δεν υπάρχει έλεγχος της ποιότητας, δεν υπάρχει έλεγχος της ακρίβειας ε, ε, των στοιχείων εντοπισμού, γεωγραφικού εντοπισμού που προκύπτουν στι και το συμπέρασμα βεβαίως στο οποίο φτάσατε είναι ανησυχητικό ότι υπάρχει ένα σημείωμα το οποίο ε, προειδοποιεί ε, για την ε, ποιότητα και τον κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ποιότητα αυτών των δεδομένων και πρέπει να υπάρχει ένα έλεγχο των ποιοτήτων όποτε αυτό είναι εφικτό. Οπότε αναρωτιέμαι, αυτέ οι διαδικασίε που θεσπίσατε, που προφανώ δεν αρκούν για να επιληθούν όλα τα προβλήματα, αυτέ οι διαδικασίε δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη-μέλη. Ακόμα και κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν τα τα δεδομένα τα ίδια, αυτά τα δικά σας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε από την υπόθεση είναι ότι τα δεδομένα των επικοινωνιών είναι ένα εργαλείο το οποίο ε, ουσιαστικά ε, σχετίζεται άμεσα, άρρηκτα με την ε, προσωπική ζωή, την ιδιωτική ζωή, την ιδιωτικότητα ε, και υπάρχουν, υπάρχει μεγάλο περιθώριο λάθους. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσεκτική χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων και τη παρακράτησής τους Ε, και απευθύνομαι στην ιδανική κυβέρνηση τώρα. Ε, αυτή η υπόθεση θα μπορούσαμε να την είχαμε προλάβει εάν δεν είχε εφαρμοστεί η ιδανική νομοθεσία για την παρακράτηση δεδομένων, διότι εδώ έχουμε παραβίαση των θεμελιών δικαιωμάτων, ε, σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Κομισιόν δηλαδή θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση απέναντι τη Δανία για την ύπαρξη αυτής της νομοθεσίας. Και έπρεπε να προταθεί ένα άλλο ευρωπαϊκό νομοθέτημα. Απευθύνομαι λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στους εκπροσώπους εδώ της δανικής κυβέρνησης Έχετε μοιραστεί τις πληροφορίες αυτές με άλλα κράτη-μέλη. Έχει υπάρξει ανάλυση της κατάστασης αλλού, όπου μπορεί να έχουν προκύψει τα ίδια προβλήματα. Λέγονται τόσα για την ασφαλή συνεργασία, αλλά εδώ μιλάμε για την ασφάλεια των ανθρώπων, ε, οι οποίοι έχουν ε, συλληφθεί ε, και εκεί δεν υπάρχει καμία συνεργασία και διαφωνώ εδώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι δεν είναι αυτό το θέμα ευρωπαϊκή αρμοδιότητας. Υπάρχει σαφέ έλλειμμα βεβαίω ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε ό,τι αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία και τη συλλογή δεδομένων και επεξεργασία του. Ε, και υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ε, μεταξύ αστυνομικών αρχών των κρατών μελών. Μπορείτε να μα εξηγήσετε λοιπόν γιατί δεν κάνατε απολύτως τίποτα μετά από αυτήν την υπόθεση που έγινε δημόσια, που δημοσιοποιήθηκε έτσι, γιατί μπορεί να φανταστεί κανείς ότι υπάρχουν και άλλες οι οποίες ε, παραμένουν άγνωστες. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος Κέρνερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι συγκλονισμένος. 32 άνθρωποι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Πώς να εμπιστευτεί κανείς το κράτος δικαίου μετά και ότι είναι σωστές οι δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι από τα πιο κομβικά, τα πιο κεντρικά ζητήματα των σχέσεων κράτους-πολίτη, γέννη. Και αυτό είναι απίστευτο, πολύ μεγάλο σφάλμα. Και πραγματικά έχω σοκαριστεί. Και με την επιπολαιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ελαφρότητα με την οποία το αντιμετωπίζει. Δυστυχώς θα επαναλάβω αυτά που είπαν και προλαλήσατες, γιατί δεν απαντήθηκαν οι ερωτήσεις και θέλω να τις ξανατονίσω. Το θέμα δεν είναι τώρα πόσοι αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω του σφάλματος, αλλά και πόσοι ενδεχομένως κυκλοφορούν ελεύθεροι ως δράστες. Και δεν μπορούμε να τους κλείσουμε στη φυλακή. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Έχετε στοιχεία πολύ συγκεκριμένα σχετικά να μας δώσετε. Όταν ήρθε εδώ η Επίτροπος, είπε ότι ε, βλέπει δυνατότητα νομοθεσίας για τη διατήρηση ε, προσωπικών δεδομένων και αποθήκευση. Για λόγους προληπτικούς. Το σκέφτεστε κι εσείς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα παραθέσω σχεδόν τον συνάλφο Μπράιερ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι απολύτως περιορισμένη η αποθήκευση και η παρακράτηση των δεδομένων, γιατί όσο περισσότερα δεδομένα συλλέγουμε, τόσο περισσότερα σφάλματα μπορεί να γίνονται και λαθροχειρίες. Φανταστείτε τι θα γίνει ε, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Είναι τελείως διαφορετική η διάσταση. Ε, ξέρετε πόσοι πολίτες και πόσες ε, ποινικέ υποθέσεις υπάρχουν στην Ευρώπη. Θέλω να μας απαντήσει ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν βγάζει συμπεράσματα για ενδεχόμενη μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε ποιο βαθμό το συζητάει με άλλα κράτη-μέλη. Έχετε ενημερώσει τα άλλα κράτη-μέλη. Έχετε εξετάσει μήπως έχουν συμβεί τα ίδια και σε άλλα κράτη-μέλη. Mr. Ο κύριος Κόφουτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, στα δανεικά. Και ε, ευχαριστώ και τους δύο ομιλητές, ε, τον κύριο Λούντ και τον κύριο και Ευχαριστώ που ήρθατε για να μας ε, εξηγήσετε αυτά τα συμβάντα. Στη Δανία ήταν, δεν ήταν συμβάντα, ήταν σκάνδαλο και ο κόσμος ξεσηκώθηκε και ανησυχεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό το σύστημα όταν έρχονται οι αρμόδιοι και μας λένε ότι έγινε λάθος και θα το διορθώσουμε. Όταν περιγράφεται τι έγινε, πραγματικά αξίζει πολύ το σεβασμό μας αυτό. Και ο υπουργό δικαιοσύνη ήρθε στην Επιτροπή μας επανειλημμένα και λογοδότησε αλλά και στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έγινε αναφορά για το, το τι συνέβη και τι πήγε στραβά. Ωραία είναι αυτά και καλά, αλλά γίνεται και άλλη συζήτηση τώρα. Για ποιο λόγο ε, κρατάμε τα δεδομένα, τα διατηρούμε, τα αποθηκεύουμε και τα χρησιμοποιούμε. Και θέλω να ρωτήσω αυτό τον αστυνομικό διευθυντή. Σε ποιο βαθμό γίνεται αυτό στην ε, Δανία, σε ποινικέ υποθέσεις, πόσο συχνά χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται γενικά, ε, είναι διαδεδομένο αυτό, τα στοιχεία της τηλεπικοινωνίας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ευρύτατα διαδεδομένο στις ποινικέ υποθέσεις. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, είναι συστηματικό, είναι συχνό, είναι κάτι το έκτακτο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δώσουμε ένα εργαλείο στα χέρια της αστυνομίας πριν αποτιμήσουμε πολιτικά τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ και πάλι. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται τώρα ο κατάλογος και ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε εδώ στο πάνελ, στο βήμα, γιατί μας μένουν ακόμη 15 λεπτά. Λοιπόν, για να ακούσουμε τις απαντήσεις από τον κύριο Λούντ, ο οποίος είναι Διευθυντή Ένωση Τεχνολογία Πληροφοριών και Πολιτική Δανία. Και κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο Βεσβάρμπερκ, ο οποίο εκπροσωπεί την Εθνική Αστυνομία τη Δανία. Αλλά ίσω θα μπορούσαμε να ακούσουμε και την Κομισιόν, αν είναι εδώ. Μήπω εν συντομία θα μπορούσατε να κάνετε κάποια σχόλια από την πλευρά τη Κομισιόν. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσα μπορώ. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την έλλειψη απάντησης ε, τη κοινοβουλευτική ερώτηση. Ζήτω συγγνώμη γι' αυτό. Είχαμε ενημερωθεί ότι θα λάβετε την απάντηση αύριο στις 22. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα θέματα είχαν κολλήσει, δεν σχετίζονται με αυτό το συγκεκριμένο θέμα αφορά το πώς ε, χειρίζεται η Κομισιόν την επεξεργασία αυτών των ερωτήσεων. Επίσης ε, και εμείς ανησυχούμε από αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει. Φυσικά ανησυχούμε ως Κομισιόν που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. Απλώς δεν πιστεύουμε ότι ως Κομισιόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες συνέπειες. Δεν είμαστε αρμόδιοι. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να εξετάσουν τα συστήματα πληροφορικής, να δουν τις διαδικασίες στο δικαστικό και στο αστυνομικό σώμα και να δουν αν σέβονται τους κανόνες προστασίας των δεδομένων. Εμείς ως Κομισιόν δεν είμαστε αρμόδιοι να ασχοληθούμε με αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση που χώρα στη Δανία. Μια άλλη παρατήρηση. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε σε νέα νομοθεσία της Κομισιόν για τη διατήρηση των δεδομένων. Η Κομισιόν δεν προετοιμάζει τώρα νέα νομοθεσία για τη διατήρηση των δεδομένων. Δεν υπάρχει απόφαση της Κομισιόν θα πρέπει να προετοιμαστεί ή να προταθεί τέτοια νομοθεσία. Μας ζήτησε πέρσι τον Ιούνιο το Συμβουλίο να προετοιμάσουμε μία μελέτη. Έτσι λοιπόν αναθέσαμε σε μια εξωτερική εταιρεία τη μελέτη αυτή και έχει ξεκινήσει αλλά δεν καταρτίζουμε νομοθεσία. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν κάτι περί αυτού. Αλλά αν στο μέλλον το πράξουμε αυτό, τότε το θέμα της ασφάλειας και της ακυριότητας και της ποιότητας των δεδομένων φυσικά θα είναι θέματα παρόντα στην νομοθεσία. Δεν θα είναι κάτι που θα το παραβλέψουμε. Και φυσικά θα εξετάσουμε πάρα πολύ στενά την υπόθεση αυτή και θα έχουμε και διδάγματα. Ένα ακόμη σχόλιο. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση της Δανίας, θα πρέπει να πούμε ότι η Δανία αντιμετώπισε αυτή την υπόθεση με τον κατάλληλο τρόπο, με ένα σοβαρό τρόπο. Αναγνώρισαν τι συνέβη και ακούσαμε όλα τα βήματα που περιέγραψαν οι Δανείοι συνάδελφοι. Έγιναν πράγματα για την αντιμετωπιστή υπόθεση αυτή. Και κάτι τελευταίο. σε σχέση με την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα κράτη-μέλη. Μιλάμε για εσφαλμένα δεδομένα. Βάσει της ε, οδηγίας της προσθήκης δεδομένων και τις χρησιμοποιητικές αρχές για το, στο άρθρο 16, ο ελεγκτής των δεδομένων ε, θα πρέπει να ενημερώσει όλους ε, τους αποδέκτες στην περίπτωση που έχουν διαβιβαστεί τα δεδομένα και αν ήταν εσφαλμένα ή κακής ποιότητας. Επομένως, υπάρχει αυτή η κακη ποιότητα. Επομένω, υπαρχει αυτη η αστυνομία της δανία να ενημερώσει άλλου παραλήπτε σε άλλα κρατημέλη τρίτες χώρες που έχουν παραλάβει τα δεδομένα αυτά. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να απαντήσουμε. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Σελούντ, καταρχήν, για να απαντήσει στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ευχαριστώ. Πιο συγκεκριμένη σε ερωτήσει ε, απευθύνονταν στη συνάδελφο από την αστυνομία. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομο λοιπόν. Προσωπικά και εγώ εξεπλάγει από αυτή την υπόθεση και είδα ότι τα δεδομένα στα οποία είχε πρόσβαση ε, αστυνομία Δηλαδή, υπήρχε αποθήκευση των δεδομένων από τους παρόχους και κάποιες φορές τα δεδομένα έρχονται σε κατέργαστες μορφές αλλά η ιδανική αστυνομία είπε ότι αυτό είναι ένα ζωτικό εργαλείο για τις αστυνομικές έρευνες. Πραγματικά λοιπόν εξεπλάγει που χειρίστηκαν τα δεδομένα με αυτόν τον μη κατάλληλο τρόπο. Φυσικά ότι έγινε έγινε. Πιστεύω ότι είναι θετικά τα βήματα που έχει πάρει η κυβέρνηση της Δανίας. Η δανική κυβέρνηση ε, έχει συμφέρον ε, να διατηρήσει την νομοθεσία περί διατήρησης των δεδομένων. Αυτό δεν είναι μυστικό και θέλει και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στα δεδομένα τηλεπικοινωνιών. Όμως παραμένει το πρόβλημα και ο κίνδυνος λαθών και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί όταν ληφθούν πρωτοβουλίες ε, για την νομοθεσία διατήρηση των δεδομένων είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριο Φίζε Βάμπερκ, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να τα πω στα αγγλικά ε, για λόγους ε, σαφήνειας. Έγιναν πολλές ερωτήσεις. Είπα και στα σχόλιά μου το εξής εξετάζουμε όλες τις υποθέσεις όπου αυτό ενδεχομένως να έχει επηρεάσει την έκβαση. Αυτή η διαδικασία είναι ακόμα εν εξελίξη. Μέχρι τώρα δεν έχω υπόψη μου καμία υπόθεση όπου ε, το σφάλμα αυτό να οδήγησε σε ε, λαθασμένη απόφαση του δικαστηρίου, σε δικαστική πλάνη. Ένα-ένα το εξεκατάζουμε με τους ανακριτές, με τους αστυνομικούς, με τους εισαγγελείς, με ειδικού για την πληροφορική και μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί καμία δικαστική απόφαση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα αν δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια. 10.700 είναι υποθέσεις. Σε καμία όμως δεν έχουμε καταλήξει ότι ήταν λάθος η απόφαση καταδικαστική. Το σφάλμα αυτό συνδέεται με το μεγάλο όγκο δεδομένο που συλλέγονται. Δεν είναι απαραίτητα ότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί και διαβιβαστεί ε, έχουν την παραμικρή ε, επίδραση στην υπόθεση. Δηλαδή από τη στιγμή που ασκείται ποινική δίωξη, σημαίνει ότι αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν τα επόμενα στάδια. Ε, δεν έχουν ληφθεί λάθος αποφάσει. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που αφέθηκαν ελεύθεροι από τις φυλακές, ε, αυτό είχε σχέση με το μορατόριο που σας περιέγραψα. Για ένα δίμηνο λήφθη η απόφαση να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα καθόλου. Δηλαδή, ε, όσοι ήταν σε κράτηση αφέθηκαν ελεύθεροι για το κράτος δικαίου και τις σωστές δικονομικές εγγύησεις. Δηλαδή, καλύτερα να τους αφήσουμε όλους ελεύθερους παρά να ε, κρατείται κάποιος αθώος. Αυτό το μορατόριο τώρα έχει έρθει και μπορούμε και πάλι να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία για να στοιχειοθετείται η δίωξη και η σύλληψη και η κράτηση. Αυτό δεν είχε να κάνει λοιπόν με λάθος αποφάσεις, αλλά ε, επειδή φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν κρατείται ως μη όφιλ. Um, additional um, Άλλες ερωτήσεις. Επιλέγω να μην απαντήσω στο θέμα του clear view. Δεν έχω τέτοια εντολή ούτε αρμοδιότητα να το σχολιάσω δυστυχώς. θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό ε, εάν ε, δεν υπήρχε απόφαση για αποθήκευση και κράτηση δεδομένων και πάλι δεν απαντώ, είναι πολιτική αυτή η απάντηση. Υπάρχουν χώρες που απευθύνθηκαν σε εμά και τις οποίες, έχουμε, τις οποίες έχουμε ενημερώσει για την κατάσταση και για το περιεχόμενο ε, των κάστοτε υποθέσεων. Απαντήσαμε σε όποιον απευθύνθηκε σε εμά και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή επιβολής του νόμου ε, έχει ενδεχομένω ερωτήσει ή αμφιβολίες, δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κύριου Κόφουτ, Κόφουτ, είναι μέχρι από το 2012. Κάθε χρόνο είναι διάφορες χιλιάδες Και αυτό αφορά φυσικά τη δίωξη σοβαρού εγκλήματο. Βαρέω εγκλήματο. Αυτά, φτάνει. Πω, πω, βλέπω δύο χέρια να σηκώνονται για να απαντήσουν. Άντε, σύντομα σα παρακαλώ όμω για να τελειώσουμε εγκαίρω. Κυρία Εντφέλτ. Ένα σύντομο ερώτημα. Είπατε ότι κοινοποιήσατε προ άλλε χώρε ότι μπορεί να μοιραστήκατε μαζί του τα δεδομένα αυτά. Να θες το ερώτημα όμως. Τώρα που γνωρίζετε ότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος Πώς, δηλαδή ε, είμαι βέβαιη ότι η δανική αστυνομία χρησιμοποιεί στοιχεία που προέρχονται από άλλες χώρες, έτσι. Θέτεται τότε το ερώτημα, πώς αξιόπιστα είναι τα στοιχεία αυτά. Μήπως τώρα ανησυχείτε κάπως. Ακούστε, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω αν μπορούμε αυτή την υπόθεση να την γενικεύσουμε σε άλλες χώρες ε, και να αφισβητήσουμε τα στοιχεία τους. Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Ε, εμείς πάντως σε σχέση με την συλλογή δεδομένων και τις υποθέσεις που επιτοπίσαμε εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε συνεργαστεί, όταν έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει συνεργασία με άλλες χώρες για τα συγκεκριμένα δεδομένα θα συνεργαστούμε μαζί τους. Όπως είπα πάντως δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα υποθέσεις όπου πάρθηκε λανθασμένη απόφαση από το δικαστήριο. Και αν κάποια στοιχεία τα έχουμε μοιραστεί με άλλο κράτος μέλος, από αυτά τα στοιχεία εννοώ, προφανώς και θα αναλάβουμε την, την απαραίτητη δράση για να αντιδράσουμε. Και πάλι εν συντομία, ε, ναι, ο κύριο Μπρέγερ, αν κατάλαβα καλά αυτό που μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι με βάση τα την απόφαση πλαίσιο για την προστασία δεδομένων υπάρχει υποχρέωση ενεργούς ε, ε ενημέρωσης για οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία ενδεχομένω να είναι λαθασμένο. Αν κατάλαβα καλά όμω, είστε σε διάλογο μόνο με τι κυβερνήσει εκείνε οι οποίε οι ίδιε ήρθαν σε επαφή μαζί σα ή έχετε αναλάβει εσεί την πρωτοβουλία να ενημερώσετε όλου του αποδέκτε αυτών των στοιχείων. Και αν δεν το έχετε κάνει, γιατί. Ακούστε. Μόνο στο βαθμό που εντοπίζουμε ε, κάποιο πρόβλημα, έτσι. Όχι επειδή απλά μοιραστήκαμε στοιχεία, πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτή τη στιγμή θα το συζητήσουμε βεβαίως κατά πόσο υπάρχει ανάγκη να κοινοποιήσουμε σε κάποιον άλλον ότι για τα συγκεκριμένα στοιχεία τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν σημασία για την εκδίκαση της υπόθεσης και πρέπει να ενημερώσουμε σχετικά. Μάλιστα, ωραία, νομίζω αρκεί για το, σημείο αυτό. Ε, ολοκληρώσαμε ακριβώς στις 5. Έχουμε ακόμα μία ώρα στη διαθεσή μας για το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Αυτό το τελευταίο σημείο σήμερα το απόγευμα ε, θα συζητηθεί και κλεισμένο το θυρών το σημείο 14. Διαπραγματεύσει για τη σύναψη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ για τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά πολιτικά στοιχεία και συνεργασία σε ποινικά ζητήματα. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε μια παρουσίαση που θα μα κάνει πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σύμφωνα με του κανόνε περί συνεδριάσεων εκκλεισμένων των θηρών, οι σύμβουλοι, οι βοηθοί, τα μέλη οι συγκητές, ε, εκπρόσωποι ε, του Προεδρίου, της, της Γραμματείας, ε, εκπρόσωποι της EDPS, του Συμβουλίου, μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα. Οι υπόλοιποι καλούνται να φύγουν. Τώρα από εκεί πέρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους ομιλητές. Ευχαριστούμε κύριε Λούντ.